είναι εγκεκριμένοι. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ αποφάσισε να ξεκινήσει διαθεσμικέ διαπραγματεύσει βάσει του άρθρου 79.4, παράγραφο 1 του ιστορικού κανονισμού. Η αντιπροσωπεία έχει εντολή για να ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα τη Ολομέλεια και ο τίτλο θα δημοσιευθεί στα πρακτικά τη σημερινή συνόδου. Βάσει του άρθρου 79.4.2, εάν ε, ένα ή περισσότεροι βουλευτέ που ξεπερνούν ε, τον αριθμό των ψήφων μέχρι αύριο μπορούν να ζητήσουν να ε, προβληθεί αντίρρηση στην έναξη των ε, διαπραγματεύσεων. Εάν δεν υπάρξει έκφραση τέτοια αντίρρηση στην Ολομέλη, η Επιτροπή ΕΚΟΝ θα ξεκινήσει τι σχετικέ